Good morning everybody. Καλημέρα. Καθίστε παρακαλώ. Πρέπει να αρχίσουμε γιατί όλοι έχουμε λυμμένες υποχρεώσεις μετά την ψηφοφορία παρακαλώ. Προετοιμάστε τις κάρτες σας ε, για την ψηφοφορία. Να αρχίσουμε με την έγκριση του σχεδίου μέρης της διάταξης. Θα ήθελα να αρχίσουμε. We'll use it. Thank you. So uh, we can start by the adoption of the agenda. Έγκριση μερίσες διάταξης πρώτα απ' όλα. Ενστάσεις. Ευχαριστώ. Μπορούμε να εγκρίνουμε και τα πρακτικά από την προηγούμενη συνεδρίαση. Ωραία. Εγκρίνονται ψηφοφορίες. Σχέδια έκθεσης για τη δημιουργία ε, ευνοϊκών όρων για την αγορά εργασίας για την ισορροπία ε, στην ιδιωτική επαγγελματική ζωή. Αποσύρθηκε η πρώτη. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 144 υπέρ κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ άρχεται Okay, so it was Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 145 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Έλεγχος άμα θέλετε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε όντως. 428 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνατε. 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 430 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 9 υπέρ κατά Αποχές ε, ε, θα χρειαστεί επαλήθευση. Έλεγχος παρακαλώ. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 9α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική η τροπολογία 230 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 228 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2.31 υπέρ, κατά, αποχές εγκρι... απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2.40 υπέρ, κατά, αποχές έλεγχος. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε η συμβαστική 15 υπέρ. Ζητώ συγγνώμη. 2.42 ξέχασα υπέρ κατά. Έλεγχος. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Ναι, απερίφθη. Η συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2.43 υπέρ, κατά, αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Όχι, όχι, διορθώνει πρόεδρος. Δε συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρας. Να περιμένουμε. εγκρίνεται. Η ε, σημαντική 22 υπέρ κατά Μην εγκρίνεται. Η 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 406 υπέρ. Α, και έχουμε και προφορική τροπολογία από θα συμπεριλαμβάνεται ήδη στην ε, τροπολογία, την ψηφίσουμε ως έχει Κατά εποχές εγκρίθηκε. Τώρα, 2.92 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. σημαντική 24. Ναι, ήταν ξεκάθαρο το αποτέλεσμα, αλλά αν θέλετε ελέγχουμε. Παρακαλώ. Για τη 292 κάνουμε τον έλεγχο. 292. 292. Απορρίπτεται. 24 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 συμβαστική πάλι. Για την 24 ζητάτε έλεγχο. Σύμφωνοι. Ψηφίστε για την 24. Να, Ναι, 25. Συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές 312 3-12 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται. Έλεγχος όμως. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Ναι, ναι, όντως απορρίπτεται. Η σημαντική 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3.17 και 3.18 ομού. Περ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται. Συμβαστική 28 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.28 και 3.29 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Είναι ξεκάθαρο. Αν θέλετε παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτονται. Ε, η συμβαστική 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Ε, εγκρίνονται. Ε, συμβαστική 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τρία τριάντα πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχος παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίθη. Συμβαστική 31. Όχι. Διορθώνει η πρόεδρος. 3.38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 344 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 347. Σωστά. Ναι, 347 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. έρχεται. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 221 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ για τη 221. Πέρας. Εγκρίθηκε. 379. Αυτή καταπίπτει. 357 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 359 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 372 και 373 ταυτόσιμες υπέρ κατά Αποχέ, απορρίπτονται. Συμβαστική 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά. Αχα. Αν είναι κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απόχέ, εγκρίθηκε. 381 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 413 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 383 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 402. Κατά τμήματα που ζητάνε οι σοσιαλιστές. Πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Το πρώτο τμήμα καταπίπτει. Και άρα ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα. Γιατί υπέρ κατά. Γιατί είναι μέσα στη συμβαστική το πρώτο τμήμα γι' αυτό. Τελευταία στιγμή την πήραμε την πληροφορία αυτή. Το ψηφίζουμε αν θέλετε και το πρώτο τμήμα για να μην υπάρξει σύγχυση. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο. Ψηφίστε παρακαλώ. Α, έλεγχος για το πρώτο. Κάποιος το ζήτησε. 402 πρώτο τμήμα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 39 κάτω 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 403 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική έλεγχος για την 43 ε, για τη 44 ήταν ξεκάθαρη η έκβαση. Ψηφίστε παρακαλώ τότε για τη 45. Για 44 θέλετε. Πέρας. Ναι. Επιβεβαιώνεται. Κρίθηκε. 4.20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγκρίθηκε. 4.21 υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. έλεγχο Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 423. Υπέρ. Συγγνώμη, διορθώνει πρόεδρο. 426 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Συμβαστική 46 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 429 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 442 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 443 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 444 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 4.45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4.59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 464 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε έλεγχος άμα θέλετε ψηφίστε ναι εγκρίθηκε τροπολογία 1 υπέρ όχι 2 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος να. Πέρασε. Ναι, απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές καταπίπτει μα περίπτει η 12 13 ναι, υπέρ κατά απορρίψαμε τη 12 και πρέπει να ψηφίσουμε τη 13 ξανά 13 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρας. Εγκρίθηκε. 22 είπε, κάτα. Αποχέ, απορρίπτα. 23 είπε, κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 26 υπέρ κατά άποχες νομίζω εγκρίνεται έλεγχος Ψηφίστε παρακαλώ. Ναι, εγκρίθηκε. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος 40 πέρασε γκρίθηκε 41 είπε Κάτω. έλεγχος παρακαλώ και για αυτή άρχεται πέρας εγκρίθηκε 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές έλεγχος 45 πέρας εγκρίθηκε συμβαστική 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά θέσεις απορρίπτεται 58 υπέρ κατά θέσεις απορρίπτεται συμβαστική 54 υπέρ κατά θέσεις εγκρίνεται συμβαστική 55 υπέρ κατά θέσεις εγκρίνεται και 56 υπέρ κατά θέσεις εγκρίνεται 79 ναι, υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρας. Εγκρίθηκε. Στα 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 57 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ την 71. Εντάξει, έλεγχος. Απορρίπτεται. 73 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται 74 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται 75 υπέρ. Κατά. αποχές... εγκρίνεται 76 υπέρ. Κατά. αποχές... 77. Έλέγχο για την 76. Όχι, εντάξει. 77 είπε. Κατά. Αποχές απορρίζεται. Η 82 είναι κατά τμήματα. Το ζήτησε το ΕΛΚ. Υπέρ. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχέ έλεγχο για το δεύτερο τμήμα τη 82. Εγκρίθηκε. Η 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ ε, κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100, 100 υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος. Εγκρίθηκε, να συγγνώμη. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτω 113 κατά τμήματα τα ζήτησε τα ECR. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1.14 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται 1.15 υπέρ. Α, κατά τμήματα. Ε, το ζήτησαν φιλελεύθερη πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, εγκρίνεται. Η 116. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ κατά αποχές ενεχώς παρακαλώ. Πέρας, εγκρίθηκε. 132 κατά τμήματα, το ζήτησε το ΕΛΚ, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές. Νομίζω επίσης εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η κυρία Φωνστόκ έχει ζητήσει το λόγο. Ναι, θα ήθελα να πω ότι σύμφωνα με το άρθρο 56.3 υπάρχει ε, ψηφοφορία μία Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε την συνεδρία της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, πρέπει να αρχίσουμε, να συνεχίσουμε μάλλον τις ψηφοφορίες. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να καλέσω όσους δεν θα συμμετάσχουν να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Ah, and my, I think that this is my Thank you. Yeah. Gut, aber Leo. Bueno, vamos a continuar. Συνεχίζουμε λοιπόν με την ψηφοφορία. Στο επόμενο σημείο της μιλησίας διατάξεως. Σχετικά με τους τρόπους που μπορεί η κοινή γεωργική πολιτική να συμβάλλει στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης ή στην Ήπεθρο της κυρίας Κιώστινγκα. Παρακαλώ, λέει η Πρόεδρος, για να ξεκινήσουμε. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά. Εποχές για να ελέγξουμε. Να κάνουμε ένα τσεκ στην 23. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Ναι, ναι, ψηφίζουμε στην 27, ξέρετε. y ε, la segunda parte con una Δεύτερο τμήμα λοιπόν με την ενσωματωμένη τροπολογία την προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά αποχές δεν είδα τίποτα 36 άρχεται η ψηφοφορία Hay tres personas que no Τρεις δεν ψήφισαν, εν πάση περιπτώσει πέρασε τις ψηφοφορίες όμως. Εγκρίνεται. Η σημαντική πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. τη 41. Άρχεται. Σε cierra la votación. Πέρας. Εγκρίθηκε. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 45 σε 3 μέρη πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές για να κάνουμε ένα τσεκ στο δεύτερο τμήμα σε φιέρα Πέρας. Απορρίφθηκε. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. 47. Σε Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 55 σε δύο τμήματα το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 5 υπέρ. Συγγνώμη λέει η πρόεδρος. Όχι. Η 1. Η τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 τώρα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15, 15 με συγχωρείτε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε στην τελική ψηφοφορία άρχεται Σε cierra la votación. Πέρας. Δεν λείπει κανεί από ό,τι βλέπω. Ξαναλέει πέρας η πρόεδρο. 26 υπέρ, 3 εποχέ, καμία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Και περνάμε στην γνωμοδότηση του κυρίου Κουρτασούν για το Ευρωπαϊκό εξάμεινο και πάμε στην ψήφο. Η τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 σε 3 τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. πέντε σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η έξι σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 1 υπέρ κατά αποχές ε, νεκρίθησαν λοιπόν οι τροπολογίες και ολοκληρώσαμε τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες.